Ε, ε, Νοεμβρίου θα ε, γίνει η επόμενη συνεδρίαση και στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα. Λύεται η συνεδρίαση.